οι ψηφοφορίες που προβλέπονται για σήμερα. Πρώτα-πρώτα έχουμε την έκθεση Σένφλτ, εξάλληψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Θα ψηφιστεί ολόκληρη η έκθεση ονομαστικά και τώρα ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Μισό λεπτό. Πέρας. Και εγκρίνεται. Έκθεση Λάγκη. όμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα. Όλοι μαζί η, έκθεση, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φίσας Αϊξελά. Συμφωνία Εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση Κολομβίας και Περού. Προσχώρηση της Κροατία. Ψηφίζουμε όλο το κείμενο. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Καβαντά ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών. Ψηφίζουμε όλο το κείμενο μαζί με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουν. Πέρασα. Εγκρίνεται. Έκθεση Άντερσον. Εξάλληψη παρανόμου εμπορίου προϊόντων καπνού όλο μαζί το κείμενο ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Φέρμπερ. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Έχουμε την τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Με ανάταση χειρός κατά αποχές εγκρίνεται η δέσμη υπαριθμών να και τώρα θα ψηφίσουν πρώτα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάταση χειρός υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Ακόμη μια έκθεση του κυρίου Φέρμπερ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων. Τροπολογία υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Με ανάταση χειρός. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η δέσμη υπαριθμών 1 και τώρα ψήφιση της Επιτροπής η πρώτη επιτροπή Ανατασχυρώσει υπέρ κατά κρίνεται το νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση στάση. Διορισμός μέλο του Ελληνικού Συνεδρίου. Κυρίου Γρημάντας Σάτζιους. Μυστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Πρέντα. Για την έκθεση του 15 Συνοχή αναπτυξιακή Πολιτικής. Μετά την παράγραφο 8 έχουμε μια προφορική τροπολογία του κυρίου Κέρντσα. Ο οποίος αν θέλει μπορεί να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ανάψε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχει ένας διαιτικός μηχανισμός ε, για, ούτως ώστε να μπορέσουν να ασχίσουν τα μέτρα Juncker για να υπάρχει μια πολιτική συνοχής και σε περίπτωση που υπάρχει δικογνωμία μεταξύ των διαφορετικών ε, πολιτικών θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνης όσον αφορά τις βασικές κατευθυντήριες και εκείνη θα κρίνει ανάλογα με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, γιατί εάν δεχθούμε αυτή την τροπολογία τότε αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ε, ε, ε, επιβεβαιώσουμε αυτή την, ε, το ψήφισμα το οποίο πήραμε το 2013. Ιδάλλως, δεν θα έχουμε ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά την συνοχή των πολιτικών μας και ιδίω όσον αφορά αυτή την προσφυγή στην διαιτησία. Ακριβώ όπω έλεγε ο παλιός συνάδελφο Μπολόνο, και έτσι θα μπορέσουμε σε περίπτωση άρνηση να οδηγηθούμε στο ότι έχουμε ε, μια πολιτική συνοχή που θα είναι σαν ένα μαχαίρι που δεν έχει λάμα. Υπάρχει κάποια ένσταση για αυτή την προφορική τροπολογία. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 40 βουλευτές οι οποίοι να ενίστανται και να σηκώνονται από τη θέση τους. Α, επομένω δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτή την προφορική τροπολογία. Οπότε πάμε στην επόμενη τροπολογία που είναι η τροπολογία υπαριθμών 1 για την παραγράφο 10. Με ανάταση τη χειροσπή είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Παράγραφος 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίζουν. Πέρας. Και εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Το πρωτότυπο κείμενο. Ανάταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά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 Παραγραφός 24. Μιλούμε για το αρχικό πρωτότυπο κείμενο. Ανάταση χειρός υπέρ, κατά, αποχές. Θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Και εγκρίνεται. Παράγραφος 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Το αρχικό πρωτοτυπο σε τρία τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 33 σε δύο τμήματα, ανάταση χειρός και εδώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές, θα γίνει επαλήθευση ηλεκτρονική, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 40 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παραγραφός 41 ανάταση χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική ε υπέρ κατά αποχές Ανάταση χειρός, παρακαλώ σαφώς να κρατάτε ψηλά τα χέρια σας, αλλιώς είναι δύσκολο. Ψηφίζουμε, πέρας. Και εγκρίνεται αιτιολογική F, ανάταση χειρός, υπέρ κατά αποχές. Και εδώ θα πρέπει να γίνει επαλήθευση. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Χόιμπουχ. Νέα συμμαχία επιστημιστική ασφάλεια και διατροφή. παράγραφο 2 σε δύο τμήματα. Το πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, να τα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Ανάταση χειρός. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος Πέντε. Έχουμε το εδάφιο μόνο 2 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 18. Ανάταση χειρός. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ανάταση χειρός. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά. Εποχές εγκρίνεται. 25 σε δύο τμήματα το πρώτο. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με ανάταση χειρό. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 28. Ανάταση χειρό. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 34 Πρώτο εδάφιο. Σε δύο τμήματα το πρώτο. Υπέρ, κατά. Α, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Εδάφιο 2. Του αρχικού κειμένου, με ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34, εδάφιο 6, ανάταση χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 36, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 59 σε δύο τμήματα. Το πρώτο ανάταση χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται παράγραφος 72. Υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονική. Τώρα ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 85. Ανάταση χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε την ιδεολογική παραγραφό 26, αρχικού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αιτιολογική 37 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αιτιολογική C του αρχικού κειμένου και εδώ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε La votazione Approvato. Και εγκρίνεται το ψήφισμα το, στο σύνολό του τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Votazione chiusa. Πέρασε. Εγκρίνεται έκθεση στο Λόγιαν, Αξιολόγηση διεθνών λογιστικών προτύπων. θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται έκθεση Φανόρντεν. Υποστήριξη της ειρήνης. Συνεργασία Ένωσης, ΟΗΕ και Αφρικανικής Ένωσης. Παραγραφός 6 του αρχικού κειμένου. Ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 σε 3 τμήματα. Το πρώτο με ανάταση χειρός. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Δυνατά στις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Το αρχικό κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται παράγραφος 22 δυνατά ισχυρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, το 8 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη 1, σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση σε καθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Υπάρχει μια τροπολογία της Επιτροπής Γεωργίας υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει τώρα Έρας εγκρίνεται Έκθεση μακιντάερ, Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράγραφος 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, διανατάς της υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8 σε δίτηματα Πρώτο τμήμα, Ανατάσσεω τη χειρό υπέρ, κατά Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές θα κάνουμε επαλήθευση ηλεκτρονική που έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20 δυνατά της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 24 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται πέρας απορρίπτεται τρίτο τμήμα πάλι με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει τώρα τέλος εγκρίνεται παράγραφος 25 και εδώ ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας εγκρίνεται Παράγραφος 27, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28. Και εδώ ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει τώρα. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 30. Ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει τώρα. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, καταπίπτει. Πάμε στην παράγραφο 32, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, διανατάς χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε επαλήθευση. Ξεκινάει. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 42. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Δυνατά στις χειρός υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, διανομαστικής ψηφοφορία. που άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφο 47. 46 οθόνη ο πρόεδρος. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 47. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφο 58 σε δύο τμήματα δυνατά στις χειρός υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 70 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα δυνατά χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 74. Πρώτο τμήμα διανομαστικής ψηφοφορίας που άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα διανομαστικής ψηφοφορίας που άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διατάσσεται χειρό υπέρ. Κατά αποχές θα κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. πέρας εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη C σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα είναι ανατάσεις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας εγκρίνεται τρίτο τμήμα διονομαστικής ψηφοφορίας άρχεται εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη γιώτα του αρχικού κειμένου, διανομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Q σε δύο τμήματα, δυνατά ισχυρό, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη R. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Δυνατά σχηρό υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συνολικό ψήφισμα διανομαστικής ψηφοφορίας που άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην έκθεση Όιτεμαν. Ενίσχυση τη καινοτομία οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της μελλοντική Ευρωπαϊκής Διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Παράγραφος 10 του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Διανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 31, δυνατά ισχυρός, χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 31, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 32, πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, Παρακαλώ σηκώνετε το χέρι σας ψηλά γιατί δεν βλέπω. Επαναλαμβάνω. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Δυνατάς χειρός. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται αλλά κάνουμε μια εξακρίβωση άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 33, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Εταιρική σκέψη α του αρχικού κειμένου, τέταρτα τμήματα, πρώτο τμήμα, εντάξει χειρό, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές θα κάνουμε έναν έλεγχο άρχεται πέρας εγκρίνεται τέταρτο τμήμα υπέρ είναι τάσος κατά αποχές εγκρίνεται τετρική σκέψη σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη D του αρχικού κειμένου, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη I σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιονική σκέψη J, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος λοιπόν για το δεύτερο τμήμα σε τη λογική σκέψη J. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Μικρή διαφορά. Το ψήφισμα τώρα στο σύνολό του διονομαστικής ψηφοφορίας άρχεται. Εγκρίνεται λοιπόν. Πέρα των ψηφοφοριών εδώ. Πάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Ενώ οι συνάδελφοι εγκαταλείπουν την αίθουσα. Ας περιμένουμε δύο λεπτά για την εκένωση της αιθούσης. Ένα λεπτό λοιπόν. Και μετά θα ξεκινήσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Πάμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Έκθεση Φέρμπερ. Η αγορά χρηματοστατικών μέσων. Συνάδελφε Πόλτσακ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.